Ζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Και τώρα ερχόμαστε εις ε, τις ε, παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού. Πρώτα η κυρία Σκριντελεύσκα από το ΕΛΚ. Κύριε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ίσια ε, ε, αμοιβή για τους άνδρες και τις γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. Πρέπει να υπάρξει ισότητα ε, στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αρχή αυτή περιέχονταν ήδη στη συνθήκη της Ρώμης. Έχουν γίνει πρόοδοι για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, αλλά οι διαφορές εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές. Ο μέσος όρος είναι 16,5% η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν υπάρχουν ε, θα, θα, δεν μπορούν να γίνουν θαύματα οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, πρέπει να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη ώστε να ακολουθούν και να εφαρμόζουν μια πιο αποτελεσματική πολιτική. Πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εφαρμόζονται καλές και βέλτιστες πρακτικές και το 2013 ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους υπάρχει τόσο περιορισμένη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Η επόμενη ε, ομιλήτρια είναι η κυρία Διέρε. Ευχαριστώ. Μέσα στα πλαίσια της ε, Παγκόσμιας ημέρας υπέρ της γυναίκας θα ήθελα να δούμε το πρώτο πρόγραμμα καινοτομίας και υπέρ της γυναίκας. Μιλάμε για το 2020 και για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε έτσι ώστε να μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες ε, αποτελούν το 30% του ερευνητικού προσωπικού και του πανεπιστημιακού. Ε, θα πρέπει λοιπόν ως Ευρωπαίοι να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το κεφάλαιό μας έτσι ώστε να προωθήσουμε την καινοτομία και την παραγωγικότητα. Εάν υπάρχει ισότητα υπάρχει μεγαλύτερη καινοτομία στην ε, κοινωνία. Θέλουμε την πλήρη συμμετοχή των γυναικών έτσι ώστε να φτάσουμε στο στους βασικούς στόχους το 2020, δηλαδή να έχουμε αριστεία στην επιστήμη χάρη στην ε, συμμετοχή των γυναικών. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μιράντα από τους Πρασίνους. Ο τομέας ε, της ναυπηγικής βρίσκεται σε ικτρή κατάσταση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη ε, Γαλλικία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με βάση τις ε, εξελίξεις στον τομέα της ναυπηγικής όπου αποσχολούνται 10.000 εργαζόμενοι. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι χάσαμε 3.500 θέσεις εργασίας και επίσης άλλες 1.000 θέσεις είναι επισφαλής. Βρισκόμαστε σε οριακή κατάσταση, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο γιατί αυτό θα είναι ολέθριο για την οικονομία της χώρας μας. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει άμεση απάντηση και να μας πει πώς θα έχουμε καλύτερη ε, δημοσιονομική πολιτική μέσα στην εξήγηση της ναπίκη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία ώστε τα μεγάλα τα μεγάλα φορτηγά να μπορούν να κυκλοφορούν στις οδούς από την πίσω, από την πίσω πόρτα με αποτέλεσμα να υπάρχει συμφόρεση και αυξανόμενα επίπεδα, επίπεδα ρήπανσης. Η Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει να αναλύσει τη διαβούλευση που μόλις ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Η ερμηνεία της Επιτροπής σε ό,τι αφορά είναι η εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων ώστε να ξεπεράσουν τα φορτηγά τη διάσταση των 25 μέτρων με δυσάρεστες συνέπειες για τους φορολογούμενους, για, τη ε, για τη συμφόρηση. Πόσες γέφυρες θα πρέπει να κατασκευαστούν ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αυτά τα γιγαντοφορτηγά λαμβάνονται μονομερείς αποφάσεις για θέματα που θα επηρεάσουν τις τοπικές περιοχές και τις τοπικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να λαμβάνονται οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις υπόψη. Ευχαριστώ κύριο Τούσας. Που υπόσχονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Η ανεργία καλπάζει με 25 εκατομμύρια ανέργους και αλματώδεις ρυθμούς επέκτασης σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει για τις γυναίκες και τους νέους όπου ένα ένας στους δύο είναι άνεργος στην ελλάδα και την ισπανία. στην ελλάδα η ανεργία εκτινάχθηκε στο 23% πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. την ίδια ώρα η κυβέρνηση στην ελλάδα από κοινού με την τρόικα προχωρούν στην κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας μειώνουν δραστικά μισθούς και συντάξεις η μείωση των μισθών των νέων κατά 32% συνοδεύεται από ε, σήμερα με τη μείωση κατά 22% του πενιχρού επιδόματος ανεργίας. Ζωή κόλαση για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Χιλιάδες νέοι παίρνουν το δρόμο της αναγκαστικής μετανάστευσης, περιπλανόμενοι στην Ευρώπη και σε άλλες υπήρους, αναζητώντας επιβίωση. Αλλά και εκεί αντιμετωπίζουν τα δουλεμπορικά γραφεία, τις ελαστικές μορφές δουλειάς, μισθούς πείνας που δεν καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες οι νέοι που ζουν ή ξεριζώνονται από την πατρίδα τους δεν πρέπει να αποδεχτούν την ανεργία τη φτώχεια και την εξαθλίωση που τους καταδικάζει η καπιταλιστική βαρβαρότητα. σε αυτές τις συνθήκες απαιτείται κοινή οργάνωση και πάλι των εργαζομένων για την προστασία και την ανακούφιση τους. Ευχαριστώ. Ο Κονίλιο Βαλάντιμ Τουντόρ έχει τώρα το λόγο. Κυρίες και κύριοι, το 1923 και 33 είχε πει δεν έχει σημασία ποιος θα ψηφίσει αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει, ε, υπάρχουν πολλές μαφίες και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία ε, μαφία δημοσκοπήσεων. Μπορώ να σας πω ότι στη Ρουμανία αυτή η κατάσταση έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις διότι οι δημοσκοπήσεις ε, στις δημοσκοπήσεις δαπανώνται ε, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει έλεγχο των δημοσκοπήσεων σε επίπεδο Ευρώπης και οι παραβαίνοντες να τιμωρούνται. Δεν μπορούμε να ζητάμε ελεύθερες εκλογές τη στιγμή που υπάρχουν ε, μεγάλες, μεγάλη μνοθεία στις δημοσκοπήσεις. Ευχαριστώ το λόγο ο κύριος Λούχαν. Αγαπητοί συναδελφοί, για πολλούς λόγους βλέπουμε ότι ε, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες και στον οικογενειακό τομέα. Δυστυχώς πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι πλήττονται άνθρωποι μέσα στα πλαίσια της οικογενειακής εστίας. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία να προβλέπουν αυτές τις καταστάσεις και να προτρέχουν αυτόν. Οι οικογένειες και μέλη της οικογένειας γίνονται θύματα, ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά θα πρέπει τα κράτη-μέλη με κοινοτικά κονδύλια να υποστηρίξουν τέτοια προγράμματα όπως το Δάφνη και να υποστηρίξουν την καταπολέμηση της οικογενειακής βίας. Δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες, γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, πολυσχηδής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Νταντσίλα. Η Ρουμανία όπως και άλλες χώρες γνώρισαν έναν δυσίωνο χειμώνα με ε, πάγο και ε, δυσίωνες καιρικέ συνθήκες. Γι' αυτό πολλοί παραγωγοί βρίσκονται σε ε, πολύ δύσκολη θέση. Στη Βράντσα 44.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν πληγεί και έχουν υποστεί ζημίες από 60-100%. Θα πρέπει λοιπόν να αποζημιωθούν οι παραγωγοί οποροκυπευτικών γιατί δεν γίνονται επαρκείς επενδύσεις θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το λάβει αυτό και να υποστηρίξει τους παραγωγούς που έχουν πληγεί και για να αναζωογονηθεί αυτός ο τομέας των οποροκυπευτικών που έχει μεγάλη σημασία και για τους καταναλωτές γιατί αυξάνονται οι τιμές των οποροκυπευτικών όταν σπανίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χρυσόγελος εκ των Πρασίνων. Πριν από λίγη ώρα συζητήσαμε εδώ για την έκθεση για την ισότητα των δύο φύλων. Αλλά θα ήθελα να πω ότι ενώ στη συζήτηση αυτή που κάνουμε εδώ μιλάμε για τη βελτίωση των θέσεων της θέσης γυναίκας στην ελλάδα τα πράγματα έχουν πάει προς τα πίσω. το σύνθημα ίση αμοιβή για ίση εργασία μοιάζει πάρα πολύ μακρινό και η ανεργία αυτά είναι πλέον σε πρωτοφανή επίδα και για τα δύο φύλλα, όμω οι επιπτώσει κρίση είναι πιο βαριέ για τι γυναίκε. Οι κοινωνικέ υποδομέ που ήταν έτσι κι αλλιώ αδύναμε στη χώρα μα ερικνώνονται, πλήττοντα κυρίω όμω τη θέση των γυναικών. Γιατί και τα δύο φύλλα ξεκίνησαν από διαφορετικέ αφετηρίε, μια και η ενεργεία των γυναικών ήταν έτσι κι αλλιώ υψηλότερη στο παρελθόν, ενώ τώρα έχει διπλασιαστεί οι γυναίκε ήταν σε καθεστώ εργασιακή απορρίθμιση πολύ πριν αυτή θεσμιστεί επισήμω. οι περικοπέ μισθών έπληξαν περισσότερο τι γυναίκε που έτσι κι αλλιώ αμείβονταν χαμηλότερα ίσω και κατά. 20%. όμω για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τη ελληνική κρίση πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μια εξορρόπηση μείωση των εισοδημάτων με στοχευμένα μέτρα βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και τη κοινωνική συνοχή αν θέλουμε να μιλάμε στοιχειοδό για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. και αυτό πρέπει να περνάει σε οποιαδήποτε μέτρα και πολιτικές Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα είναι Σχούμπερ. Ευχαριστώ. Η συμφωνία μεταξύ Τρόικας Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Πορτογαλίας δείχνει ότι πλήττεται ο πορτογαλικός λαός. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση οικονομικής ανέχειας. Έχουμε χάσει 157.000 θέσεις εργασίας. Φτάσαμε στο 20,3% δίκτυ ανεργίας. Βρισκόμαστε στο κατόφλι της ανέχειας. Υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία εισοδημάτων και κατανομή εισοδήματος. Δυστυχώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δυσίωνη θέση. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει υποστήριξη του τομέα υγείας. Αυτό είναι οδυνηρό, διότι υπάρχει και υψηλή θνησιμότητα στην Πορτογαλία. Η κυβέρνηση όμως και το Σοσιαλιστικό Κόμμα προβάλλουν τις ίδιες αξιώσεις. Θα πρέπει όμως να ανακτήσουμε τους στρατηγικούς τομείς και να φτάσουμε σε μία σωστή ε, οικονομική αναζωογόνηση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νούνο Μέλο. Ευχαριστώ. Η Πορτογαλία ζει περίοδο μεγάλης ε, ξηρασίας το 30% της επιφάνειας βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης ξηρασίας, ενώ ένα 70% σε κατάσταση μερικής ξηρασίας. Αυξάνεται το κόστος ενέργειας, το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται και αυξάνονται και οι τιμές των προϊόντων. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη των Ευρωπαίων. Κάνω μια έκκληση προς τα θεσμικά όργανα έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και η υπερθέρμανση του πλανήτη που πλήττει τις χώρες του νότου της Ευρώπης τα πλαίσια της ΚΑΠ και των ειδικών μηχανισμών υπέρ της γεωργίας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γιάννε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χτες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια ε, της μεγαλύτερης τρομοκρατικής βίας κατά της Ευρώπης στη Μαδρίτη την 11η του Τρίτου του 4. Είχαμε πολλά θύματα, ιδιαίτερα στη Μαδρίτη. παρά τις έρευνες που διενεργήθηκαν και παρά τους θανάτους είδαμε ότι δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την τομοκρατία. Ούτε το Λονδίνο το κατάφερε, ούτε η Αμερική. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε την αξιοπρέπεια και την θέληση των θυμάτων. Η Πιλάρ Μανχών έχασε το παιδί της ένα νέο 20 ετών και ε, προέβη στην σύσταση οργάνωσης υπέρ των θυμάτων και των οικογενειών τους και υποστήριξε αυτόν τον θεσμό με μεγάλη αξιοπρέπεια και καρτερία. Το λόγο έχει ο κύριος Κουμουτσάκος. Η αναδίπλωση η αναδιάρθρωση ε, του ελληνικού χρέους με τη μεγαλύτερη στην ιστορία ανταλλαγή κρατικών ομολόγων είναι πια γεγονό. είναι μια μεγάλη αναπνοή αλλά μία μόνο σε έναν επώδυνο μαραθώνιο με δρομέα τον ελληνικό λαό που υφίσταται δραματικές θυσίες και μεγάλες προσπάθειες. η ελληνική οικονομία διασχίζει μια έρημο λαο που υφισταται δραματικες θυσιες και μεγαλες προσπαθειε η ελληνική κοινωνία μια ερημο υφεση η ελληνικη κοινωνια μια ερημο ανεργια και το εμπόριο διασχίζει μια έρημο λουκέτων η ελλάδα χρειάζεται επιγόντως μια όαση μια όαση ανάπτυξης. έως τώρα στη χώρα μου εφαρμόστηκε το παράδειγμα και το πείραμα της σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας. τώρα ταυτόχρονα πρέπει να εφαρμοστεί και το παράδειγμα της ανάπτυξης. γι' αυτό χρειάζονται νέες και εφαρμόσιμες ιδέες. η συγκρότηση μιας ελληνοευρωπαϊκής αναπτυξιακής τράπεζας είναι μια σοβαρή και ρεαλιστική ιδέα την πρότεινε πρόσφατα ο αρχηγός του κόμματός μου στη γερμανίδα καγκελάριο. πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να την στηρίξει και να την προωθήσει. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κουσκέρη. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στο 2012-5002 που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα όπου αναλύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν δεθεί, δοθεί στην αεροπορική εταιρεία Air Malta με αποτέλεσμα να επηρεαστούν δυσμενώς οι πτήσεις και οι μετακινήσεις. Όλοι ανησυχούν για το μέλλον τους. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του ΑΕΠ της Μάλτας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μια μείωση 1.300 υπαλλήλων από την ΕΡ Μάλτα, ενώ δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για αυτή την κατάσταση. Η λύση για την κρίση δεν θα έπρεπε να είναι η καταπίεση των εργαζόμενων μια κατάλληλη σύνδεση ανάμεσα στη Μάλτα και διεθνείς προορισμούς είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομίας και για τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων, νέων θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών στη Μάλτα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κούσμπη. Ευχαριστώ. Αυτό τον τελευταίο καιρό είχαμε διάφορες πληροφορίες στην Ευρώπη σχετικά με το τι κάνει το κόμμα ελευθερίας και ο αρχηγός του ο κύριος Βίλντερ στην Ολλανδία και οδήγησε σε προσφυγές ε, κατά των ξένων οι πρώτοι οι οποίοι ε, κατηγορούνται είναι οι Πολωνοί που εργάζονται νόμιμα σε Ολλανδικές εταιρείες και θεωρούν ότι ε, ε, υφαρπάζουν τις ε, θέσεις Ολλανδών εργαζομένων. Σύμφωνα με τις Ολλανδικές τράπεζες οι Πολωνοί καλύπτουν το 2,3% του ΑΕΠ και πολλοί πρέσβεις έχουν επέμβει. Εν τω μεταξύ ο κύριος Βίλντερς λέει ασχοληθείτε εσείς με τα δικά σας και ε, εκπλήσωμε ότι ο Πρωθυπουργό δεν, ε, ε, δεν τοποθετείται και θα έπρεπε να μπορέσει να λάβει θέση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πελάγιο Ροντρίγκε τώρα έχει το λόγο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στις ε, περικοπές ε, τις ε, δημοσιονομικές που πλήττουν το σύστημα υγείας σε πολλές χώρες. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές για τα ερευνητικά προγράμματα. Και αυτό το βλέπουμε και στην Καστίγια Λαμάντσα. Βλέπουμε ότι γίνονται εξετάσεις, μάλλον ε, απαλήφονται εξετάσεις ιδιαίτερα στα νεογέννητα. Στα νεογέννητα για να δούμε πώς εξελίσσεται, πώς έχει το γένομά τους και να ανοιχνευθούν ασθένειες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εγγυηθούμε αυτή την αρρωγή και το δικαίωμα στην υγεία. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να μην ε, κόβουμε προγράμματα ιδιαίτερα στον τομέα της νοσοκομιακής αρρωγής. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ναβιντέλοβα. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που η κυρία Βασιλείου είναι εδώ γιατί θέλω να, γνωρίσω, να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει τώρα η ανεργία των νέων που ανέφερε και ο κύριος Μπαρόζο είναι κάτι που χρειάζεται να επέμβουμε και να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα κατά της ανεργίας πρέπει να στηρίξουμε και την επιμόρφωση και αυτό γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, το βλέπουμε άλλωστε και από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό όμως το οποίο δεν βλέπουμε είναι μια ιδέα που δεν ε, υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τι δεξιότητες θα χρειαστούμε στο μέλλον ποια θα είναι η κατεύθυνση την οποία θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ποια πορεία θα ακολουθήσει και θα έπρεπε να υπάρξει μια συζήτηση με εμπειρογνώμονες από τον εκπαιδευτικό χώρο, από τη βιομηχανία για να δούμε ποιες είναι οι δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον για να μην επανέλθουμε στα προβλήματα του παρελθόντος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριος Κούτας. Αγαπητοί συνέδελφοι, θα πρέπει να προστατεύσουμε την πνευματική διοκτησία στα πλαίσια της ΑΚΤΑ και νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο η ε, άκτα είναι το κατάλληλο μέσο. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή προασπίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Σύμφωνα με το ΔΕΚ ε, υπάρχουν και άλλα μέσα η αποδοτικότητα της άκτα είναι περιορισμένη, διότι η παραποίηση δεν αντιμετωπίζεται με το άκτα κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να υπογράψουμε, να κυρώσουμε ένα κείμενο το οποίο να υπερβαίνει τα πλαίσια της άκτα μέσω και της Παγκόσμιας ε, Οργάνωσης Εμπορίου εκτός ΠΟΕ η άκτα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτα. Ευχαριστώ Κύριε Σταμπόιντι. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ε, μου δίνετε για πρώτη φορά το λόγο σαν ε, πρόεδρος και είναι ε, ένα ερωτηματικό αν θα πρέπει και τα κράτη να τιμωρούνται εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσω αφαιρέσεως των πόρων συνοχής. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις, οι κοινότητες δεν πρέπει να τιμωρούνται και αυτή η μη ύπαρξη ε, κυρώσεων ε, δεν είναι σωστή ε, διότι βλέπουμε ότι αφαιρέθηκαν 500, 500 εκατομμύρια ευρώ από τους ε, Ούγγρους ε, ε, ενώ δεν έγινε κάτι παρεμφερές για τους Ισπανούς οπότε αύριο πρέπει να δούμε τι θα αποφασιστεί και θα υπάρχει μεγαλύτερη σοφία από ό,τι παρελθόν Ευχαριστώ Η κυρία Ιρυγκογιάν Περέθ έχει το λόγο τώρα Ευχαριστώ να σας επισύρω την προσοχή στον Σημερινό όπου υπάρχει δικτατορία από το 79 εδώ και 20 χρόνια καταδιώκει το μόνο δημοκρατικό κόμμα στη 9 του μηνός ο Βεσεσλάου Μασόκο ε, βρίσκεται υποκράτηση και δεν ξέρουμε πότε θα απελευθερωθεί. Έτσι η διεθνής κοινότητα, η UNESCO δηλαδή, δεν μπορεί να δεχτεί 3 εκατομμύρια δολάρια για να τιμήσει με αυτό το έπαθλο ένα δικτάτορα. Θα θέλαμε λοιπόν να μην ξεπληθεί η εικόνα του ε, δικτάτορα αυτού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 20% των παιδιών πεθαίνουν πριν από τα 5 τα πέντε τους χρόνια. Θα πρέπει να ζητήσουμε ελευθερία και να ζητήσουμε και την απελευθέρωση του Βενσεσλάου λόγω. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοστέλο έχει τώρα το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει κατά πόσο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πώληση φαρμάκων για τους οποίους χρειάζεται, χρειάζεται συνταγογράφηση αλλά που αγοράζονται χωρίς συνταγή ε, σε χώρες, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στους δρόμους του Δουβλίνου. Αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αϊπνίας πολλούνται στους δρόμους του Δουβλίνου και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα εάν τα πάρει κανείς σε συνδυασμό με ενόπνευμα ή άλλες ουσίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαθεσιμότητά τους οφείλεται στην κρίση την οικονομική που μαστίζει την Ιρλανδία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το πόσο μπορεί να ληφθεί η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της πώληση ε, φαρμάκων χωρίς ε, συνταγογράφηση στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Σάρμπο έχει το λόγο. Το ίμιση του πληθυσμού της ε, Ρουμανίας βρίσκεται σε κατάσταση ανέχειας. Δυστυχώς όμως ε, δεν μπορεί το κράτος να βοηθήσει μέσω ε, του τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, καθώς και η διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει πελατιοκρατία και να μην δράει η μαφία του κυβερνώντος κόμματος θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αν βγούμε από την κατάσταση λιτότητας όπου δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν με τα ψυχία μισθών με τα οποία ζουν. Σας ευχαριστώ. Köszönöm szépen. Áttérünk Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της μερισίας διατάξεως, δηλαδή την έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ σχετικά με